Καλησπέρα σας. Καθίστε παρακαλώ πολύ. Είμαστε ελάχιστοι. Χαίρομαι πάντως που εκπροσωπούνται οι πολιτικές ομάδες, οι περισσότερες. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θα φτάσουν σε λίγο. Είναι Δευτέρα άλλωστε, η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας. στα τελικά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε ευθύ αμέσω με την ε, έγκριση της μερίσιας διάταξης. Πρώτο σημείο. Μπορούμε να εγκρίνουμε την μερίσια διάταξη, εκτός αν υπάρχουν βέβαια αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Και όσον αφορά το σημείο 2, έκριση των πρακτικών της συνεδρίασης των 17-18 Φεβρουαρίου θεωρούνται και τα πρακτικά ότι εγκρίνονται αν μέχρι το τέλος της ημέρας δεν έχουμε αντιρρήσεις ή τροποποίησεις για τις ανακοινώσεις. Μία ανακοίνωση ενδιαφέρουσα θεωρώ στις 16 Μαρτίου, δηλαδή σε δύο ημέρες το πρωί, στις 10 η ώρα το πρωί, θα έχουμε μία συνάντηση όπου προσεκλήθην οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει να κάνει με, τον, με το EUMED, με το δίκτυο των πανεπιστημίων δηλαδή των, της Μεσογείου και με τον κύριο Παντσέρη, ο οποίος είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες Μαγκρέμπ. Η Μαρία Τερέζα Χιμένες Βερμπάτ επίσης θα είναι παρούσα και θέμα συζήτηση θα είναι η συνεργασία στον τομέα τη επιστήμης μέσω του δικτύου αυτών των πανεπιστημίων τη Μεσογείου. Νομίζω ότι ε, στη συνάντηση αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, έχουμε και ένα δικό μα ψήφισμα με το οποίο συμφωνεί και το υπόλοιπο κοινοβούλιο εφόσον εγκρίθηκε το Νοέμβριο και είχαμε πει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και φοιτητών που ε, συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο Πανεπιστημίου της Μεσογείου και θα πρέπει να γνωρίσουμε επίσης ότι ακόμα και φοιτητές πρόσφυγες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο δίκτυο αυτό. Πρόκειται λοιπόν να έχουμε στις 16 Μαρτίου έχουμε τη συνάντηση αυτή με τρία πανεπιστήμια της Ιταλίας τα οποία θα υποδεχθούν 50 φοιτητές πρόσφυγες. Ελπίζω και άλλα πανεπιστήμια να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό και έστειλα μια επιστολή και στον Αβρατσίς, και στην κυρία Μογκερίνη προκειμένου πραγματικά να ακολουθηθεί το παράδειγμα αυτό και από άλλα πανεπιστήμια. Έχει πάρει λοιπόν η επιστολή αυτή σε διάφορου πρίτανε διαφόρων πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ κάθε πανεπιστήμιο λειτουργεί αυτόνομα και εντελώ ανεξάρτητα. Είναι καλό όμω να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερα πανεπιστήμια προκειμένου να υποδεχθούν φοιτητέ πρόσφυγε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική η συνάντηση αυτή που θα έχουμε σε δύο μέρε. Γλωσσικό καθεστώ. Estone, Lituano, Πολάκο, Sloveno, Bulgaro ή Rumeno. Ε, ε, Υπάρχει δερμήνια προφανώ και στα ελληνικά. Μεταδίδεται μέσω web streaming η συνάντηση. Απόφαση των συντονιστών της 18ης Φεβρουαρίου. Το κείμενο έχει αποστελεί σε όλους και νομίζω ότι εγκρίνεται τα συμπράσματα αυτά καθότι δεν υπήρχαν καθόλου αντιρρήσεις. Επίσης, τα εγγραφά σας θα δείτε μία σύντομη παρουσίαση της αποστολής που κάναμε στο Πίλσεν της Τσεχίας που χώρα τον Νοέμβριο 2015 και προτού περάσουμε στην πρώτη έκθεση για την οποία η γήτρια, γνωμοδότηση μάλλον, να προσθέσω κάτι ακόμα. Μετά τις επαφές που είχαμε με τον Επίτροπο Ναύρατσιτς στην τελευταία μας συνάντηση, στα πλαίσια της Επιτροπής μας, έστειλα μία επιστολή στον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς καθότι δεν δόθηκε ικανοποιητική απάντηση από τον πρόεδρο Γιούνκερ. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Σούλτσα έστειλε μια άλλη επιστολή Γιούγκερ. στη συνεχεια ο προεδρος σουλτσα αφορά την, το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2018. Ξέρετε ότι με το ζήτημα αυτό ασχολήθηκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η Ιταλική Προεδρία και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική πρωτεύουσα και το πολιτιστικό έτος 2018. Ξέρετε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, αλλά το ζήτημα έχουν θίξει και διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης για ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως το γνωρίζετε, ζήτημα το οποίο έθιξε και πριν από λίγο και που έχει να κάνει με την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Απασχόλησης με θέμα πρόσφυγες, κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Αποφασίσαμε και πολύ σωστά με τους συντονιστές να γνωμοδοτήσουμε ως Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού. Ζητήσαμε δηλαδή να μπορούμε να μπλακούμε περισσότερο καθότι θεωρώ ότι η πτυχή του πολιτισμού και της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντική και για την προσφυγική κρίση και για το προσφυγικό ζήτημα. καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Απασχόλησης. Η δική μας η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει όμως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό. Και επιμένουμε σε ζητήματα όπως η κατάρτιση, η διαδίου μάθηση και η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα των προσφύγων. Προτού προχωρήσω στην ανάλυση της γνωμοδότησης αυτής, πρέπει να σας πω ότι στις 21 Μαρτίου 12 το μεσημέρι θα είναι καταληκτική η ημερομηνία για τις τροπολογίες. 26 Απριλίου η ψηφοφορία σε εμά και στις 25 Μαρτίου θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ξέρετε ότι πρέπει να επιρρεωζόμαστε σε πολύ σύντομα κείμενα πλέον συγνωμοδοτήσεις. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση για το προσφυγικό ζήτημα. Εξ αρχής λοιπόν θέτουμε το ζήτημα της ενσωμάτωσης και της ένταξης ακόμα και όσον αφορά τον τομέα της παιδείας Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνικονομική ένταξη των προσφύγων και ότι η πτυχή του πολιτισμού και της παιδείας είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνία. Δεν, δεν μπορώ να ακούσω την αγγλική διερμηνία. Ακούω μια άλλη γλώσσα στο αγγλικό κανάλι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αγγλική διερμηνία. Καταφέρατε να με ακούσετε ή δεν ακούσετε τίποτα. Ωραία. Σα έλεγα λοιπόν ότι στη γνωμοδότηση αυτή προσπάθησα να αναφερθώ σε κάποιε προτεραιότητε. Η πρώτη προτεραιότητα είναι μια ολιστική σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση και τη ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω του πολύ σημαντικού ρόλου που δραματίζει η πρόσβαση στην παιδεία και η πρόσβαση στον πολιτισμό. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντική προπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των προσφύγων και ιδίω για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εκμετάλλευση και προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε μια κάποια προοπτική στι οικογένειε οι οποίε επενδύουν στα παιδιά αυτά και προκειμένου να έχουμε και μια γλωσσική και πολιτιστική διαμεσολάβηση. Και επίση θα πρέπει να προωθηθούν και κάποιε πρωτοβουλίε όπω να δημιουργηθούν συγκεκριμένε πλατφόρμε προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευση για τα παιδιά αυτά, τα οποία θα πρέπει να μπορούν και αυτά να πηγαίνουν στο σχολείο. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μα απασχόλησε και στο ψήφισμα που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το οποίο ασκούμε πολύ μεγάλη πίεση είναι να αυξηθεί η ποσόστοση της χρηματοδότησης η οποία θα πρέπει να δίνεται στην ανθρωπιστική βοήθεια για το έτος 2016 κατά τη διάρκεια δηλαδή της παραμονής των προσφύγων στους διάφορους καταβλισμούς για παράδειγμα θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν απαραίτητη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση από το συνολικό προπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 30 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον προβλέπονται για το 2016 χάρη εν μέρη και στην δική μας συμβολή και συμβολή της Επιτροπής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο του 2016 στα πλαίσια παιδί της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου Κορυφής. Κάτι εξίσου σημαντικό είναι ο πολιτιστικός, διαπολιτισμικός, διαθρησκευτικός διάλογος, η διαβίου μάθηση, η πολιτική και την νεολαία και τον αθλητισμό, καθώς επίσης Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Θέλουμε να προωθήσουμε επίση πρωτοβουλίε υπέρ τη συνεργασία μεταξύ όχι μόνο των δημοσίων αρχών των κρατών μελών, αλλά και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ίδιων των κοινοτήτων των προσφύγων, πολλέ φορέ ε, προσπαθούν με έναν τρόπο πάρα πολύ άμεσο να προωθήσουν την καλύτερη πρόσβαση των προσφύγων στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό να αφαιρθούμε επίσης και σε κάποιες ε, αρχικές πρωτοβουλίες που έχει κάνει αρκετά διστακτικές αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Plus. Πάλι και εκεί προβλέπονται κάποια σχέδια ενσωμάτωσης και ένταξη των προσφύγων. Και πάλι στα πλαίσια των προγράμμων αυτών υπάρχουν οι απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι. Σε καμία περίπτωση, και το είπαμε αυτό και στον Επίτροπο Ναύρατση, δεν ζητούμε επιπλέον πόρου αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για το έτο 2016. Από το 2017 και μετά θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε περισσότερου πόρου, ακόμα και από το περιθώριο ευελιξία που προβλέπει ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κάτι ακόμα Αναφερόμαστε και σε μία ακόμα πρωτοβουλία, γίνεται μία σαφής αναφορά στη γνωμοδότησή μου στους περίφημους εκπαιδευτικούς διαδρόμους, στους οποίους ανεφέθηκα και πριν από λίγο και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει και στη συνδιάσκεψη που θα έχουμε μεθαύριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συνεργασία της UNIMED, να καταφέρουμε δηλαδή να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και της Ένωσης Μεσογειακών Πανεπιστημίων, της UNIMED δηλαδή. Αυτά κατάφερα να εντάξω στην γνωμοδότηση αυτή. Ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένο ο αριθμό των λέξεων που μπορούμε να έχουμε σε γνωμοδοτήσει. Αυτό είναι το πρώτο μου σχέδιο. Προσβλέπω όμω και στην δική σα συνεισφορά και στι δικέ σα παρατηρήσει. Η Πέτρα έχει πρώτη το λόγο. Ja, Σε ευχαριστούμε πολύ ε, ένα πολύ καλό σχέδιο νομοδότηση, ε, το οποίο θεωρώ πραγματικά ποιοτικό. Θα ήθελα απλά να κάνω ένα σχόλιο, ε, το οποίο έρχεται στη συνέχεια τη τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Επιτροπό Ναρβαζίτση. Δηλαδή, είχα πει ότι σε κάθε περίπτωση η Επίτροπη θα πρέπει να ξεκινήσει τον αναπροσανατολισμό, αν θέλετε, του Erasmus ε, Plus και να αρχίσουν κάποια κονδύλια από αυτό το κομμάτι να απορροφούνται από το τομέα τη διαχείριση του ε, ε, προβλήματος ε, με του πρόσφυγε. Για παράδειγμα, μα είχε πει ο Επίτροπος ότι ήθελε κάποια από αυτά τα κοντήρα να κατευθυνθούν για παράδειγμα προς, την, προς γλωσσική γλωσσικής εκμάθησης για τους πρόσφυγες αλλά του εξήγησα ότι δεν είναι ο στόχος αυτός του Erasmus Plus δεν είναι για αυτόν τον λόγο δεσμευμένα αυτά τα κοντήλα και η Επιτροπή δεν μπορεί αυτόνομα αν θέλετε μόνο μερός να ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο τους στόχους τους οποίους έχουμε ορίσει για το Erasmus Plus. Ε, νομίζω κάτι τέτοιο είναι πολύ επικίνδυνο. Όλοι μας αναγνωρίζουμε την αξία του Erasmus Plus ε, ε, και βλέπουμε βέβαια κάθε χρόνο ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα projects που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και χρηματοδοτούμε λιγότερα ακριβώς γιατί είναι περιορισμένοι και οι πόροι. Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο ότι δηλαδή όλα όσα θα λάβουν χώρα στο επίπεδο της διαχείρισης του προσβητικού προβλήματος συμπεριλαμβανομένων και των ε, πρωτοβουλειών για την γλωσσική εκμάθηση και γενικά συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλειών για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών δεν μπορούν αυτά τα κονδύλια να προέλθουν από τα όσα έχουν ήδη δεσμευθεί για τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένω να βρεθούμε αντιμέτωποι με την ε, κατηγορία ότι ξέρετε τι κάνατε, ε, πήρατε τα χρήματα του Εράσμου σε και προσπαθήσατε τώρα να χρηματοδοτήσετε και άλλα ζητήματα. Πέραν δηλαδή των, ε, των στόχων Δηλαδή το ότι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε πολιτισμικού χαρακτήρα ε, project με το Εράσμο, προφανώ και θέλουμε να το κάνουμε, αλλά ε, χρηματοδότηση γλωσσικών σεμιναρίων για πρόσφυγε, όχι πραγματικά κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στου στόχου του Εράσμου και ενδεχομένω θα πρέπει να το ε, θέσουμε και ρητά, δηλαδή να το διευκρινίσουμε μέσα σε αυτό εδώ το κείμενό μα. Δηλαδή προφανώ πολιτισμικό διάλογο είναι κάτι που μα ενδιαφέρει, ναι κοινωνική ένταξη, ναι και στην κοινωνική ένταξη και βέβαια εδώ θα αναφερόμουν γενικότερα στην κοινωνική ένταξη ανθρώπων ευάλωτον, αλλά από εκεί και μετά όταν αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους ε, μέτρα, δηλαδή ε, ε, πρωτοβουλίες γλωσσικής εκμάθησης για πρόσφυγες, όχι δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εχθεί στους στόχους του Erasmus ΣΥΝ. Ας το θέσουμε λοιπόν εδώ, ρητά, Οπότε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι στο μέλλον, για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι μέλλον με, την, με τις κατηγορίες που σας ανέφερα μόλις τώρα δηλαδή να μας πούνε αύριο μεθαύριο ότι ε, τελικά δεν αναφέρατε κάτι τέτοιο στη δική σας νομοδότηση. Συμφωνώ με την ησυχία σας, θα το διευκρινίσουμε. Σεράιν παρακαλώ. Ναι, οι αγρότες ε, τελικά έχουν μπλοκάρει ε, περισσότερα από όσα νομίζαμε, γι' αυτό άργησα λίγο. Ο κύριος ε, Μαλίνο, δυστυχώς ο, ο δεν κατάφερε να βρεθεί σήμερα εδώ μαζί μας, οπότε θα ήθελα να διαβάσω μια δήλωση από την πλευρά του Στιώδους και θα ήθελα να πει το εξή, ότι ο αριθμό των προσφύγων και των μεταναστών στα κράτη-μέλη έχει αυξηθεί πρωτόγνωρα. Ε, και το ΕΛΚΕ χαιρετίζει την ε, ατζέντα τη Επιτροπή για τη Μετανάστευση που κάνει μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και να βρει και μέσω πρόθεσμο και μακροπρόθεσμη λύση όπω ε, καλύτερον έλεγχο των συνόρων, καλύτερη οργάνωση από κοινού με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του συστήματο του Δουβλίνου και ε, με, με σκοπό βέβαια να εφαρμοστούν σωστά αυτά τα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα παραμείνει, ε, θα, θα διατηρήσει τον ηγετικό τη ρόλο στον τομέα τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί βέβαια μετανάστε θα χρειαστεί να επιστρέψουν στι χώρε του επειδή είναι οικονομικοί μετανάστε. Ωστόσο κάποιοι πρόσφυγε ούτω ή άλλω θα επιστρέψουν από μόνοι του στι πατρίδε του όταν θα τελειώσει η ένοπλη σύραξη. Κάποιοι από, αυτού ενδεχομένω να αποφασίσουν να παραμείνουν μαζί μα εδώ μαζί με τα παιδιά του και θα πρέπει να διασφαλίσουν την πρόσβαση ε, στην ε, ε, εκπαίδευση των, αυτών των γενών οι οποίε είναι πιο ευάλωτε και ε, και για παράδειγμα στο, επίπεδο, στο, στο, στο πλαίσιο της επιστροφής τους στις χώρες τους ή σε περίπτωση παραμονή τους εδώ. Ε, και προφανώς είναι δύσκολο στο πλαίσιο και τις παιδιές να ε, ενθαλαχθούν και οι ε, αξίες της χώρας υποδοχές. Γι' αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι προσπάθειες της εκπαίδευσης. Δηλαδή το να διαχειριστούμε τα σημερινά προβλήματα είναι σημαντικό για να βρούμε μια λύση για το μέλλον. Στη διαφορετική περίπτωση απλά να βάλουμε την κρίση για την επαύριο και η, ε, η ένταξη στην αγορά εργασία σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρχει αναγνώριση των επαγγελματικών ε, δεξιοτήτων οι οποίε ε, αναγνωρίζονται από, από, το, από τη χώρα υποδοχή. Η αναγνώριση λοιπόν των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσόντων, η επαγγελματική κατάρτιση προφανώ θα πρέπει να αναγνωρίζονται όπω και ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταδίκη του κάθε είδου ε, ξενοφοβία και μεσολοδοξία και προφανώ θα πρέπει να γίνουν και προσπάθειε ε, ε, εντατική γνωστή εκμάθηση και προετοιμασία για την συμμετοχή στο κανονικό σχολικό σύστημα. Ο κ. Ζεμαρινόφ θεωρεί λοιπόν πω το σχέδιο γνωμοδότηση είναι πολύ καλοσορροπημένο προ τη διατύπωσή του, αλλά θα βάλει κάποιε τροπολογίε για να διευκρινιστούν τα εξή. Καταρχήν, καλό ορισμό των ετούντων άσυλο και προσφύγων στο πλαίσιο τη γνωμοδότηση τη ΚΑΛΤ. Επίση, η παιδεία ω βασικό σημαντικό στοιχείο της κοινωνική ένταξη και ένταξη στην αγορά εργασία. Τρίτο στοιχείο, ο σημαντικός ρόλος των στοχευμένων μέτρων εκπαίδευση και επενδυματική κατάρτισης για διαφορετικέ ομάδες ε, προσφύγων και ε, υποστήριξη ε, των εκπαιδευτών και των δασκάλων ε, που υποστηρίζονται τους πρόφυγες. Νομίζω πως ο Σκιώδης εδώ αναφέρει ε, πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά όπως είπε και η συνάδελφος ε, Κάμαρβερντε, δεν μπορούμε μέσω των υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για παράδειγμα μέσω του Erasmus Plus, να χρηματοδοτήσουμε άλλες, άλλου χαρακτήρα πρωτοβουλία. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να προέλθει από τους προπολογισμού των κατομελών αλλά και άλλων μεγαλύτερων ταμείων, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ταμεία τα οποία είναι αρμόδια για μέτρα και καταλληλότερα για μέτρα όπως αυτά της κοινωνικής ένταξης. Ούτως ή ο κλάδος ε, της ε, παιδείας ε, πάντοτε έχει πρόβλημα υποχρηματοδότησης. Οπότε αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε για παράδειγμα διασυνοριακή ανταλλαγή δασκάλων ή ανταλλαγή πληροφοριών και μαθητών Προφανώ μπορούμε να το κάνουμε, αλλά και για παράδειγμα ένταξη μέσω του αθλητικών δραστηριοτήτων, για παράδειγμα και σε ε, διεθνέ επίπεδο, κάτι τέτοιο και όλε αυτέ οι δραστηριότητε έχουν και κάποια, κάποιο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη, αλλά να λέμε ότι θα ε, χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα τέτοιε δραστηριότητε μόνο από τα δικά μα κονδύλια όπω το Erasmus Plus, προφανώ δεν είναι σωστό γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει και σε νέε συζητήσει στα ίδια τα κράτη-μέλη ε, και θα ε, θα, θα θέσουμε δηλαδή επιτάπητος και νέα, ε, ε, νέα ζητήματα σε ό,τι αφορά το, το ζήτημα του προσφύγων, οπότε τα εφιστάμενα κονδύλια θα πρέπει να παραμένουν δεσμευμένα για τους αρχικού του στόχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Λίουερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Ίσως δεν θα σας εκπλήξει πάρα πολλοί συνάδελφοι αν σας πω πως το σχέδιο γνωμοδότησης δεν ευθυγραμμίζεται με πολλές από τις απόψεις της δικής μου ομάδας. Ο κύριος Τζαμπάσκι είναι ο σκιώδης εισηγητής, αλλά όπως μας είπε η, η, και η Σαμπίν είναι αρκετοί συνάδελφοι που λείπουν. Θα τον εκπροσωπήσω λοιπόν εγώ εδώ. Ο αριθμός των προσφύγων αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστιος και η πολιτική ενσωμάτωση θα μπορούσε να προσφέρει κάτι, αλλά θα πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να σχεδιαστεί από πριν, έτσι ώστε να μην έχουμε καθόλου κατασπατάληση πόρων ή χρόνου. Άρα χρειάζεται να αναλύσουμε το ποιοι είναι, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι πολλές φορές, πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία μας, εάν θέλουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, τι επαγγέλλονται, ε, έχουν τη δυνατότητα να μάθουν την γλώσσα της χώρας οικοδεσπότε πότε και πολλές ακόμα ερωτήσεις πριν δώσουμε μια απάντηση σωστή στο πρόβλημα αυτό ή εν πάση που να προσεγγίζει αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε στην παράγραφο 3 προτείνεται και μάλιστα αρκετά επίμονα να διπλασιάσουμε τα κονδύλια για την παιδεία και για τις επίγουσες δράσεις στα κράτη-μέλη. Αυτό ίσως δεν ευθυγραμμίζεται με τις εθνικές πεπιθήσεις και αυτή η έκκληση για νέους πόρους ε, αμφισβητείται γιατί ερωτώ εγώ από πού θα προέρχονται αυτά τα κονδύλια η φορολογία ε, ήδη είναι πάρα πολύ υψηλή και το Εράσμους ΣΥΝ νομίζω ότι σχολιάστηκε πολύ ε, σωστά ο κίνδυνος που ελοχεύει από τους συναδέλφους τώρα εγώ είμαι συντανιστή και στην Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη για την ομάδα μου και ξέρετε πω για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη δεν ε, θέλουν ε, να ασχολούνται ε, όσοι δεν είναι αρμόδιοι με αυτά τα δύο ταμεία και νομίζω ότι θα εξακολουθούν να πιέσουν προ αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για τι κοινέ αξίε, για του ετούντε άσυλο και του πρόσφυγε στην Ευρώπη, ποιε είναι αυτέ οι κοινέ αξίε, δεν τι ορίζουμε κάπου. Και τέλο, θα έπρεπε άρα για τα κράτη-μέλη στα πανεπιστημία τους να έχουν κάποιους διαδρόμους πανεπιστημιακούς οι οποίοι ε, θα αφορούν τους πρόσφυγες, μα δεν είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας και πού θα οδηγήσει σε ποσοστώσεις για τους, προσφυγές, για τους πρόσφυγες σε κάθε πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αυτά λοιπόν γενικά σίγουρα θα ακολουθήσουν τροπολογίες και περιμένουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε. Θα σας απαντήσω μετά. Βίλτε, παρακαλώ. You are shadow, Σκιώδης δεν είστε. Νόμιζα ότι ήσασταν σκιώδης. Φανταζόμουν ότι θα θέλετε το λόγο. Δεν ζητήσετε το λόγο. Μόργαν λοιπόν. Κι εγώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ε, συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Όπως είπατε πολύ σωστά κυρία Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε εδώ πέρα να δούμε πόσα στοιχεία μπορούμε να εντάξουμε σε ένα κείμενο το οποίο σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να είναι αρκετά ευσύνοπτο. Το σχέδιο γνωμοδότησης, το σχέδιο έκθεσης μάλλον έχει να κάνει με τους πρόσφυγες και οι περισσότεροι συνάδελφοι είπαν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν περαιτέρω μέτρα από αυτά τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο έκθεσης. Πάντως η δική μας γνωμοδότηση δεν έχει να κάνει απλώς με τους πρόσφυγες, αλλά έχει να κάνει με την ενσωμάτωσή τους και με τη χρησιμοποίηση πολιτιστικών μέσων. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε εκ των προτέρων να λέμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε περισσότερα μέσα ή ότι θέλουμε να του αποκλείσουμε. Νομίζω ότι στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε μια συζήτηση πιο στρατηγικής φύσης όσον αφορά το ζήτημα του προπολογισμού και των μελλοντικών περικοπών και όχι μόνο για το έτος 2017. Αναφέρουμε προφανώς το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη του στις μελλοντικές τουλάχιστον ενδείξεις που θα δώσει πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μια νέα κρίση, μια έκτακτη κρίση όπως η προσφυγική κρίση. Είναι πολύ δύσκολο να μην καταφέρουμε να πάρουμε πόρους από άλλα ταμεία ή από άλλες πολιτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούμε να ανακαταμείνουμε κάπως τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και την κρίση αυτή. Πάντως νομίζω ότι στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης θα μας δοθεί δυνατότητα να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση. Μάρεγκαλ παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Και μόνο για να μοιραστώ μαζί σας και το πνεύμα αλλά και το γράμμα αυτής της γνωμοδότησης. Διαβάζοντας τη γνωμοδότηση λοιπόν, έχω κάποιες ιδέες που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, κάποια στοιχεία για να προσθέσουμε, όχι γιατί έχω αντιρρήσεις, κάθε άλλο να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα. Ίσως χρειάζεται μια αναφορά στην ε, αναθεώρηση ε, του Πουδουπού έτσι ώστε και η εκπαίδευση και, και ο πολιτισμός να λάβουν υπόψη την ένταξη των προσφύγων στις κοινωνίες μας. Και δεύτερον, που συνδέεται με την παρατήρηση που μόλις έκανα. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε απερίφραστα και γραπτά πως όλες οι δαπάνες, όλοι οι πόροι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι η καλύτερη δυνατόν επένδυση που μπορεί να κάνει η Ευρώπη γιατί θα κερδίσουμε φίλους, θα δημιουργήσουμε γέφυρες προς το μέλλον, θα συνεισφέρουμε σε μια μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ κοινωνιών είναι η πιο κερδοφόρα επένδυση από όπου και να το δει Και μία λεπτομέρεια ακόμα για τα θέματα παιδείας, για το κατά πόσο θα πρέπει αυτή η ένταξη να γίνεται και στα συστήματα παιδείας ε, χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις και χωρίς να χρησιμοποιηθούν και να δημιουργηθούν ε, παράλληλες δομές. και για να παρουσιάζονται στα δικά μας σχολεία, στα δικά μας πανεπιστήμια, στα δικά μας ΤΕΙ. Γιατί έτσι κι αλλιώς στη δουλειά και στο επάγγελμα θα σταθούν δίπλα μας. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά. Ο κύριος Βέρα. Υπάρχει ε, ο κίνδυνος τον οποίο γνωρίζουμε όλοι να δημιουργηθούν εδώ παράλληλες ε, κοινωνίες. Ε, γι' αυτό θα ήθελα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο να αναπτύξουμε ολιστικές στρατηγικές σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και γενικότερα την παιδεία των μεταναστών. Όμως βέβαια όλες αυτές οι προσπάθειες εξαρτώνται στο σύνολό τους από τη χρηματοδότηση. Ε, μία λοιπόν ε, εναλλακτική είναι να διαθέσουμε περαιτέρω κονδύλια, συμπληρωματικά κονδύλια για τέτοιου είδους ε, ε, ε πρωτοβουλίες και μία δεύτερη. και βέβαια σε σχέση με αυτό είναι δύσκολο να διασφαλίσουμε συμπληρωματικά κονδύλια όπως ακούσαμε μόλις τώρα ε, συμπληρωματικά κονδύλια και το τομέα της ε, ε, παιδείας. Ίσως όμως θα μπορούσαμε να βρούμε εδώ μια λύση, δηλαδή στα, στους σχολικούς αν θέλετε προϋπολογισμούς των κρατών μελών υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση αυτής της παιδείας των μεταναστών. Δεν γνωρίζω δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την πλήρη ένταξη των μεταναστών αν δεν λάβουμε υπόψη μας αυτή την πτυχή της εκπαίδευσης και της κουλτούρας ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Δεν μπορούμε δηλαδή να χάνουμε σε καμία περίπτωση χρόνο σε σχέση ακριβώς με ε, την εκπαίδευση των παιδιών. Όμως, όπως είπε ότι ο προηγούμενος ομιλητής, ε, ε, ε ενδεχομένως οι, τα corridors όπως έχουν προταθεί δεν μπορούν να αποτελέσουν μακροπρόθεσμα λύση, ίσως για μία περίοδο, ναι. Ε, για παράδειγμα για να αποκτηθούν οι βασικές γλωσσικές δεξιότητες. Όμως ε, σε διαφορετική περίπτωση με τη δημιουργία τέτοιων κόρδων θα δημιουργήσουμε διαφορετικές παράλληλες κοινωνίες όπως είπα, πράγμα που φυσικά δεν μπορεί να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Ja, eine ganz Ναι, απλώς να κάνω μια διευκρίνηση, Πρόεδρε, για να μην υπάρξουν παρανοήσεις. Προφανώς αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και υποχρέωση του κρατών μελών να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στι ευθύνε του, να καλύπτουν δηλαδή τι υφιστάμενε ανάγκε, να παράγουν δηλαδή την κατάλληλη, ε, να παρέσουν την κατάλληλη σχολική εκπαίδευση και να ενσωματώσουν και τέτοιου είδου πρωτοβουλίε ένταξη δηλαδή μέσα στα σχολικά του συστήματα. Νομίζω πως ε, αυτή η υποχρέωση, αυτό το καθήκον δεν μπορεί ούτως ή άλλως να το αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κονδύλια μας δεν επαρκούν για κάτι τέτοιο, αλλά κάτι τέτοιο υπερβαίνει και τις αρμοδιότητες μας κατά πολύ, σε σχέση δηλαδή με αυτές που αναφέρονται στις συνθήκες. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη, να δημιουργήσουν για παράδειγμα τέτοιου είδους ε, σχολικές τάξεις χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή ε, μεθόδους για την καλύτερη ένταξη των παιδιωτών μεταναστών. Αυτό που μπορούμε εμείς ενεργά να κάνουμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμπληρωματικά on the top αν θέλετε προγράμματα, για παράδειγμα σε επίπεδο διαπολιτισμικών projects και ούτω καθεξής. Εκεί σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια τόσο του Erasmus Plus όσο και του ε, Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe. Ε, εκείνο που νομίζω πως ήδη έχει αποφασιστεί είναι ότι η ανθρωπιστική βοήθεια η οποία απευθύνεται σε καταβλισμούς ε, προσφύγων οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα στην Ιορδανία ε, και στη Λιβύη, αυτά λοιπόν ε, τα κονδύλια θα πρέπει να επενδυθεί και στην εκπαίδευση των παιδιών τα οποία ακριβώς βρίσκονται σε αυτούς τους προσφυγικούς καταβλισμούς. Αυτό είναι ε, ε, σημαντικό και αναφέρεται και μέσα στην έκθεση γιατί πρόκειται για κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα οποία δηλαδή έχουμε και εμεί ε, λόγο. Από εκεί και μετά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλώ να επιθύνουμε μία έκκληση στα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν τέτοιου είδου πρωτοβουλίε στα σχολικά του συστήματα, στου σχολικού του προπολογισμού και από εκεί και μετά αυτό που μπορούμε εμείς να συμπληρώσουμε κάποια διαπολιτισμικά προγράμματα. Όμως δεν μπορούμε να αναλάβουμε ένα καθήκον, ε, μια αρμοδιότητα η οποία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και αυτό νομίζω ε, συμπεριλαμβάνει και σεμινάρια για παράδειγμα ε, γλωσσικής εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής τέτοιου είδου, ε, για παράδειγμα, προγράμματα είναι αρμοδιότητα του κρατών μελών. Γενικά, η πολιτική στον τομέα τη παιδεία είναι εθνική αρμοδιότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πολύ σύντομα, ε, αύριο η κυρία Γκαριάτσο, αφού στο πλαίσιο τη ακρόαση θα επιστρέψει πιο λεπτόμερο στα όσα εμεί προετοιμάζουμε από την πλευρά τη Επιτροπή μα. Η Πρόεδρο είπε ότι ε, μέχρι στιγμής ήμασταν λίγο αργοί, αν θέλετε, δεν ήταν τόσο ταχύς η δική μας ε, ρυθμή. Όμως ε, για τα τέλη του Απριλίου εμείς όπως γνωρίζετε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντα για την μετανάστευση ετοιμάζουμε και κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά την νόμιμη μετανάστευση εκεί περιλαμβάνεται και ένα σχέδιο κοινωνικής ένταξης των μεταναστών που έχει προετοιμαστεί από κοινό από τις διάφορες συναρμόδιες ε, ε, μόναδες της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και θα αποφασιστεί ποια ακριβώ στοιχεία του θα συμπεριληφθούν, γιατί βέβαια μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση περιλαμβάνει διαφορετικού χαρακτήρα ε, ε, ε, ε τομεί. Αλλά βέβαια οι ε, Επίτροποι θα αποφασίσουν τελικά ποια ακριβώ κομμάτια αυτή τη ένταξη θα περιληφθούν στην ατζέντα. Τώρα, πιο γενικά σε ό,τι αφορά τις προτάσεις τις οποίες κάνετε στο δικό σας έγγραφο και τη γενική σας προσέγγιση μπορούμε να την υποστηρίξουμε ειδικότερο το σημείο 7 σε ό,τι αφορά το Γιούνι με την Ένωση δηλαδή των Πανεπιστημίων της ε, Μεσογείου και τη δημιουργία των Corridors θα συναντηθούμε και με τον κ. Κώστα, δηλαδή τον ε, πρόεδρο της Ένωσης και θα κάνουμε ε, και μια συζήτηση για να δούμε κατά πόσο μπορούμε, μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία ω τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σχετική πρόταση συνεργασία και ποια όχι. Ε, σίγουρα εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, τους εκπαιδευτικούς ε, φορείς να υποστηρίζουν τους πρόσφυγες οι οποίες έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή και απευθείας πώς μπορούν να τους βοηθήσουν αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εκείνους τουλάχιστον οι οποίοι αποσκοπούν στο να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ε, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη τέτοιε πρωτοβουλίε έχουν ξεκινήσει και έχουν τρέξει καλά σε διάφορα κρατημέλη. Και αύριο θα ακούσετε περισσότερο, όπω σα είπα, στην ακρόαση από την πλευρά τη κυρία ε, Γκαριάτσου Και σε πολιτικό επίπεδο, όπω σα είπα, τέλη Απριλίου θα έχετε κάτι από το Κολέγιο Πλέον των Επιτρόπων. Ευχαριστούμε πολύ. Όντω, αύριο έχουμε τη συνάντηση αυτή που είναι πολύ σημαντική. Όντω, είναι πολύ πλοκό το ζήτημα και το δείχνουν αυτό και οι παρεμβάσει σα. Θεωρώ ότι ε, ορισμένες ιδέες είναι πραγματικά πολύ σημαντικές και έχουν με τον έναν άλλο τρόπο αναπτυχθεί στη γνωμοδότηση. Θα πρέπει να αποσαφανιστούν λίγο περισσότερο όμως. Κατά πρώτο λόγο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αναφερόμαστε εδώ πέρα σε πρόσφυγες. Άρα πρέπει να βασιστούμε σε αυτή την πολύ σημαντική προϋπόθεση που θέτει η Επιτροπή Απασχόλησης με την έκθεσή της, πρόσφυγες, κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά το ζήτημα της ενσωμάτωσης, το λέω και στην γνωμοδότησή μου, ότι υπάρχει αυτός ο έκτακτος χαρακτήρας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να γίνει κάτι, αλλά και από την άλλη πρέπει να συνεχίσει και μετά την πάροδο της έκτακτης αυτής περίοδου να συνεχιστούν οι προσπάθειες ενσωμάτωσης των προσφύγων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχαμε πει και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα υποδοχής και ενσωμάτωσης των προσφύγων. Πρότυπα τα οποία να είναι αποδεκτά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και που να σέβονται όμως και την αυτονομία των εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη παρατήρηση αυτή λοιπόν. Δεύτερον, το ζήτημα των ανηλίκων. Και εδώ πέρα το ζήτημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά και να προασπίσουμε την αξιοπρέπεια των παιδιών ακόμα και στα πλαίσια της Σύμβασης Προστασίας των Προσφύγων, ξέρετε ότι ακόμα και ένα παιδί, μόλον ότι δεν αναγνωρίζεται διεθνώς ως πρόσφυγας, έχει απόλυτο δικαίωμα προάσπισης και προστασίας και δυστυχώς το τομέα αυτό αυτή τη στιγμή οπισθοδρομούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανήλικοι λοιπόν θα πρέπει να μπορούν να εντάσσονται στο σχολικό περιβάλλον ανεξάρτητα από όταν έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη βασική αυτή νομική αρχή. Και κάτι ακόμα. Εγώ, όντως, κάνω μια πάρα πολύ σημαντική αμνία, αναφέρθηκε σε αυτό και ο Κάμε, η κυρία Κάμεβέρτ και ο Άντριου Λιούερ. Αναφέρομαι σε χρηματοδότηση, αλλά όχι σε επιπλέον χρηματοδότηση. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας τα 32 εκατομμύρια δηλαδή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 2% του ποσού αυτού πηγαίνει προς τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προς την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα διάφορα στρατό, στα διάφορους, στους διάφορους καταβλισμούς προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν στη γνωμοδότηση είναι ότι θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, ότι αυτό το 2% του προπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να αυξηθεί και ότι θα πρέπει η απόφαση αυτή να ληφθεί στα πλαίσια της, και της έκτακτης κρίσης που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και γενικότερα στα πλαίσια της πολιτικής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Πολλοί επίσης, η Πέτρα, η Σαμπίν και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο Erasmus Plus και σε άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπατε ότι δεν μπορούμε να αντλήσουμε πόρους από τα προγράμματα αυτά για συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, για παράδειγμα απέναντι στους ε, ενηλίκους, όσον αφορά την εκμάθηση της ε, γλώσσας της χώρας υποδοχής. Πρέπει όμως να πω και απευθύνομαι και στην Πέτρα ότι προβλέπεται στα πλαίσια του Εράσμους να δίνονται χρηματοδοτήσεις προς συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη πολιτιστικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων μη κυβερνητικών οργανώσεων, ακόμα και για την προτεραιότητα αυτή, την εκμάθηση δηλαδή της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ε, το Erasmus Plus θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει κάποια στιγμή τέτοιες ε, πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης και ένταξης. Προβλέπετε όμως. Ξέρετε ότι το ζήτημα αυτό με έχει απασχολήσει και στη δική μου την περιφέρεια, όπου έχουμε ένα, έχουμε το περιφερειακό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής μου. Ακόμα και εκεί προβλέπεται ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε πρωτοβουλίες υπέρ των προσφύγων. Σε τοπικό λοιπόν και περιφερειακό επίπεδο προβλέπεται ήδη κάτι τέτοιο. Και ο Μόργαν και ο Σβέρ είπαν ότι ε, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προβλεφθεί το αίτημα αυτό που ήδη έχει υποβάλει το Κοινοβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι σε σχέση με τη νέα αυτή επίγουσα κατάσταση που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να προβλέπονται πόροι οι οποίοι να προσανατολίζονται για την υποστήριξη των προσφύγων και να έχουν να κάνουν με το γενικότερο θεματολόγιο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ε, μετανάστευση και ότι δεν θα πρέπει να θυγούν, βέβαια τα υφιστάμενα προγράμματα. Συμφωνώ με αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνει μια διαφορετική ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την περίοδο 2017-2020 στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ένα σχετικό λοιπόν αίτημα πρέπει να υποβληθεί αυτή τη φορά από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις αυτές. Προφανώς αποσαφηνίζουν πολύ περισσότερο το κείμενό μου και θα λάβω όλες αυτές τις παρατηρήσεις πολύ σοβαρά υπόψη μου. Περνάω στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης για το οποίο συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο κύριος Στρογεύσκη τον οποίο είχα δει πριν από λίγο βέβαια και έχει ως θέμα την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του πολιτου δημοσιονομικου δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 η συμβολή του Κοινοβουλίου ενώπιση της πρότασης Επιτροπής. Θα έχουμε εδώ πέρα μια έκθεση πρωτοβουλίας από την Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώς θα πρέπει να αναμορφωθεί αυτό το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε. Είστε λοιπόν εσείς κύριε Στρογεύσκη ο συντάκτης γνωμοδότησης και σας δίνω αυτής αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω εισαγωγικά ότι δεν θα σας διαβάσω το σχέδιο αυτής της γνωμοδοτησής μου αφού το έχετε και μπροστά σας οπότε απλώ θα σα ε, παρουσιάσω ε, τα πιο σημαντικά ε, σημεία του όπως αυτά συζητήθηκαν ούτως ή άλλως. Έχουμε τρία προβλήματα τα οποία εμφανίζονται ξανά και ξανά και στα οποία θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Καταρχήν, πρόκειται για το ζήτημα των πληρωμών. Ξανά και ξανά έχουμε προσπαθήσει να το επιλύσουμε, αλλά εμφανίζεται στη συνέχεια και πάλι. Ε, το ζητούμενο δηλαδή είναι να ε, υπάρχουν ε, λιγότερα υπόλοιπα προς καθάριση και ειδικότερα σε ό,τι αφορά χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων παιδείας. Μετά, δεύτερο ζήτημα είναι ειδικότερα τα προγράμματα της εκπαίδευσης και, το Erasmus Plus. Εμείς λοιπόν ως Επιτροπή εκπαίδευση και Πολιτισμού προφανώς υποστηρίζουμε ε, ξανά και ξανά αυτό το πρόγραμμα, ε, ποιου στόχου μπορούμε να επιτύχουμε με αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, δηλαδή να τονίζουμε τη μεγάλη του σημασία. Τρίτον, ε, συχνά σε πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα τη ε, ε, αυξημένης υψηλότητας δηλαδή ανεργίας των νέων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας ώστε να μειώσουμε τα ποσοστά ανεργία των νέων. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι ο πολιτισμός ε, και η παιδεία, αυτά τα ζητήματα πολιτικής ε, δεν ε, εμπίπτουν στο τομέα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά από την πλευρά μας, ό,τι κάνουμε θα πρέπει να είναι σημαντικό και να έχει την κατάλληλη πρικοδότηση χρηματοδοτικά. Επίσης, εκείνο που αναφέρουμε σε αυτό το σχέδιο νομοδότηση είναι το πόσο, σημαντικά, ε, πόσο σημαντικές είναι οι ε, επαγγελματικές δεξιότητες ε, για προσώτα γιατί αυτά διασφαλίζουν βέβαια και την υψηλότερη απασχολησιμότητα και εδώ για παράδειγμα προγράμματα όπως το συνδέοντα στην Ευρώπη, το, η Ευρώπη για, για τους πολίτες είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπογραμμίζουμε λοιπόν την μεγάλη σημασία αυτών των project και το, την ανάγκη ύπαρξής τους και συνέχισής τους και στο μέλλον. Κάτι ακόμα συχνά στι συνεδριάσεις τη Επιτροπής μας λέμε πόσο σημαντικό είναι ο διαθρησκευτικό διάλογος για να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα όπως για παράδειγμα της ε, έλλειψης ανοχής τη ε, ε, μεσαλλοδοξία, τη έλλειψης αν θέλετε ενό ενός ανοιχτού χαρακτήρα της κοινωνίας και εκεί λοιπόν όταν θίγουμε αυτά τα ζητήματα λέμε ότι ο πολιτισμός είναι ο καλύτερος ε, τρόπος για να ξεκινήσουμε μια συμφιλίωση εδώ και εδώ ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται ο σκεφτικός διάλογος. Ε, επιτρέψτε με Ε, να πω εδώ ότι καθώς έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης για την διάμεση αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, να πούμε πως οι επενδύσεις βέβαια στο νέο, στη νέα χρονική συγκυρία είναι δύσκολότερε. Έτσι λοιπόν από το 2014 θα πρέπει ε, οι μηχανισμοί ευελιξίας για τη χρηματοδότηση που είχαμε μέχρι τώρα να ε, ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή τα κράτη-μέλη τα οποία ε, επιθυμούν να ε, συμμετάσχουν σε ένα ε, πρόγραμμα να είναι ευκολότερο να το πράξουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, την συνάδελφο η οποία είχε πάρει τον λόγο στο πλαίσιο της προηγούμενης συζήτησης και είπε ότι τα προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης δεν εντάσσονται στους στόχους του Erasmus+. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θεωρώ ότι όντω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε, ότι θα πρέπει να γίνει μια επαλήθευση όλων αυτών των προγραμμάτων. Μόργανο, Πρώτο ομιλητής και οι υπόλοιποι σκιώδει ηγητέ στη συνέχεια, Έλγα Τρούπελ και ο Άντριου Λιούερ. Καταρχά σα ευχαριστώ πολύ. Καταρχά να πω συγχαρητήρια στον συντάκτη γνωμοδότηση, τον κύριο Στρογέσκη, για την εξαιρετική αυτή ε, γνωμοδότηση που μας παρουσίασε σήμερα. Η γνωμοδότηση αυτή είναι αρκετά σύντομη όπως προβλέπεται και από τον κανονισμό, αλλά παρόλα αυτά προβλέπει και περιέχει πάρα πολλά από τα χαρακτηριστικά του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Ιδίω βέβαια επικεντρώνεται στην αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν σε διάφορα σημεία να καταφέρω να καταθέσω κάποιες ε, συγγνώμη, τροπολογίες προκειμένου να καταφέρουμε να ε, ε, περάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε κάποια σημεία, ιδίως όσον αφορά κάποια προγράμματα τα οποία αναφέρονται στην γνωμοδότηση αυτή. Νομίζω ότι Πολλές φορές έχουμε προβλήματα, όπως είπε και ο εισηγητής, με την αρχική φάση κάποιων προγραμμάτων, αλλά για κάποια προγράμματα υπάρχουν και διαρθρωτικά προβλήματα. Ιδίως όσον αφορά το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Ξέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Οριστικοποιείται αυτή τη στιγμή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα πρέπει οι πρώτες πρωτοβουλίες ήδη από το καλοκαίρι να μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Όσον αφορά τώρα το Erasmus Plus, το λέω τώρα, το, λέω και στο, το είχα πει και στο παρελθόν, ότι πολλές φορές ο τομέας νεότητας του προγράμματος αυτού έχει κάποια προγράμματα προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή κάποιων μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων. Πολλές φορές δεν διατίθενται απαραίτητοι πόροι σε εθνικό επίπεδο ή πολλές φορές οι πόροι αυτοί είναι πάρα πολύ περιορισμένοι και δεν καταφέρουν να καλύψουν τις ανάγκες συγχρηματοδότησης. Εν τέλει, όσον αφορά το πρόγραμμα Ευρώπη των πολιτών, εδώ η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ χαμηλή, φοβάμαι, για ένα πρόγραμμα το οποίο υποτίθεται ότι βρίσκεται στο κέντρο της ε, αρχής της εθνικής της ευρωπαϊκής υπηκότητας. Πέρα από τα προγράμματα αυτά Γίνεται και κάποιες συναφορές όσον αφορά την εγγύηση για τους νέους. Νομίζω ότι και για το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να υπάρχει πλήρης υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να προβλεφθεί και μια αναθεώρηση των χρηματοδοτήσεων. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο περισσότερο με τις συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν ε, ανάμεσα στο, σχέδιο Juncker, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επαναφέρουμε κάποια από τα χρηματοδοτικά κονδύλια του ορίζοντα 2020. Θεωρώ ότι τα δύο αυτά προγράμματα αλλοσυνδέονται και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσω των προγραμμάτων αυτών να τονίσουμε τις νέες πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει μέσω του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου να θέσουμε και τις βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταφέρουμε τελικά να αυξήσουμε τόσο τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και τις πιστώσεις πληρωμών. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αποκριθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις. Και αναφέρομαι εδώ πέρα και στο ζήτημα εκείνο των εκκρεμών λογαριασμών των κοντιλίων εκείνων που είχαν προβληθεί στα πλαίσια των πιστώσεων ανάληψη υποχρεώσεων, αλλά ουδέποτε τελικά δόθηκαν στα κράτη-μέλη, ουδέποτε αποτέλεσαν αντικείμενο χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτό θα είχε βοηθήσει κάπως και την προσφυγική κρίση αυτή τη στιγμή. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλοί ε, πόροι που δεν έχουν ακόμα καταβληθεί, μόλον ότι είχε προβληθεί η χρησιμοποίησή του. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και λίγο περισσότερο γενικότερα στα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ενσωμάτωση των προσφύγων. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα στα πλαίσια της Δημιουργικής Ευρώπης δημοσιεύθηκε μία πρόσκληση υποβολής προτάσεων και ξέρετε ότι θα έχουμε σύντομα και μία ακρόαση όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Ο Επίτροπος Ναυραβέτης μας είπε πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα προβλέπεται μια σφαιρική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα έχει στο κέντρο της το ζήτημα της ενσωμάτωσης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι φύγει το ζήτημα αυτό και στην τελευταία παράγραφο ο εισηγητή μας. Νομίζω ότι μέσω κάποιων τροπολογιών θα μπορούσαμε να αποσαφηνίσουμε περισσότερο το σημείο αυτό και να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται και μία αναφορά στο ότι βρισκόμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 500 εκατομμυρίων πολιτών και θα πρέπει να προωθούμε τελικά μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πολιτών αυτών. Ευχαριστούμε πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, ας είστε πιο σύντομοι στις ε, παρεμβάσεις σας. Οι επόμενοι μιλητές, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για τις προσπάθειες που έχει κάνει για αυτή τη γνωμοδότηση. Όπως μπορείτε να φανταστείτε έγινα σκιώδης και εγώ στην ομάδα μου για αυτή την ε, γνωμοδότηση. Το ε, κομμάτι ε, το πρώτο που μας ανησυχεί που είναι οι πληρωμές αυτές που αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι του προπολογισμού. Αυτό που ρωτώ εγώ είναι τα 7 χρόνια σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αλλάζει είναι σωστό επειδή κάνουμε μία αναθεώρηση ε, κάθε δύο χρόνια, ίσως εκεί αυτό θα έπρεπε να εξεταστεί. Στη δεύτερη παράγραφο δεν μπορώ να συμφωνήσω με, το, με αυτή την έκκληση να συνεχίσει αυτή η πρωτοβουλία. Ε, ξέρω πως ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια, αλλά νομίζω πως είναι ανεύθυνο να κάνουμε κάτι τέτοιο πριν την έκθεση αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα εκδοθεί την επόμενο μήνα. Και δεν έχουμε δει ακόμα πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η πολιτική για τους νέους. Οπότε ε, δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει προσφέρει κάποια αξία και όταν λάβουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως υπάρχει πειρασμός και από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως η δική τους ε, πρωτοβουλία ήταν πετυχημένη. Τώρα για τον Horizon 2020 και για το Connecting Europe εμείς μαζί με άλλες πολιτικές ομάδες ζητήσαμε ε, να ε, καταπολεμήσουμε ε, την ε, πρόθεση πόρων σε άλλα, σε άλλα προγράμματα και νομίζω ότι έχει απόλυτα δίκιο ο που ζητά να μην γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αφαιρεθούν άλλα κονδύλια από το, από το Horizon 2020 για την παιδεία και για τον πολιτισμό και τα σχετικά προγράμματα, για την ενδιάμεση αναθεώρηση, ας τη δούμε σαν μια ευκαιρία για να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα και το κατά πόσο ε, τα προγράμματα αυτά έχουν αποτελεσματικότητα για το Europe for Citizens για παράδειγμα. Επικουρικότητα μήπως χρειάζεται να ενταχθεί και αυτό στην καλύτερη νομοθεσία και στο θεματολόγιο εκεί, έτσι ώστε να μην αυξάνουμε τους πόρους χωρίς να έχουμε τα τεκμήρια που μας οδηγούν σε κάτι τέτοιο. Ένα μόνο μικρό κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, λένε κάποιοι. Αλλά τι σημαίνει αυτό δεν χρειάζεται να είμαστε επιτελεσματικοί γιατί είμαστε, είναι λίγα. Εγώ όταν ήμουνα στο Δήμο του Ντάρμπι έρχονταν οι πυροσβέστες και μου λέγανε μα είμαστε το 2% του προπολογισμού για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται το δικό μας προπολογισμό να τον περικόψετε που η παιδεία ας πούμε το 35% και πάντα υπάρχει αυτό το επιχείρημα το οποίο εγώ ποτέ δεν δέχτηκα. Τώρα για τις καθυστερημένες ε, πληρωμές και τις ε, ε, τον προγραμματισμό αυτών βεβαίως και να, ε, να αποφεύγονται γιατί θίγεται έτσι και η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οι δικαιούχοι δικαιώς παραπονιόνται οπότε εμείς δεχόμαστε τα, αυτές τις παρατηρήσεις αλλά θέλουμε και έναν αποτελεσματικό προϋπολογισμό ε, που θα δώσει τα, πίσω τα κυρίαρχα δικαιώματα στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν εφόσον αυτά παραμείνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο και θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με, το να το απευθύνω κάποιες ευχαριστίες για τα όσα προετοιμάσαι. Εμείς πάντα ε, επαγρυπνούμε για να αποφεύγουν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάζουν κάθε τόσο τον προϋπολογισμό για το θέμα της ε, ενσωμάτωσης των αλλοδαπών και των προσφύγων. Νομίζω για το προηγούμενο σημείο σίγουρα αυτό θα επηρεάσει και τα μεγάλα προγράμματα όπως το Erasmus Plus, το Creative Europe, το Europe for Citizens και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει μόνο να εξασφαλίσουμε πως θα αποφύγουμε προβλήματα με τις πληρωμές αλλά πως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια αυτών των προοπτικών να αυξήσουμε το μερίδιο αυτών των προγραμμάτων γιατί επίγει ανάγκη να χρησιμοποιηθούν έχουμε εκεί πεδίο δόξας λαμπρό. Μέσω του Euro for Citizens για παράδειγμα για πολιτισμικός διάλογος και όλα τα συναφή. Αυτή είναι η προσέγγιση μας για την αναθεώρηση, δηλαδή μια πιο εύκολη εφαρμογή των προγραμμάτων Έχουμε επικριθεί για το γεγονός ότι δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί εδώ. Ε, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη και το θέμα της ενσωμάτησης των προσφύγων είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. προτού δώσω το λόγο πάλι στο στακτή νομοδότης. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Όχι, άρα ας ακούσουμε πάλι τον εισηγητή. E, e, Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για τις παρατηρήσεις που έκαναν και τα ενθαρρυντικά τους λόγια. Προφανώς ε, θα αξιοποιήσω την δυνατότητα που έχω για να ενισχύσω ε, τα επιχειρήματα που ήδη αναφέρω μέσα στο έγγραφο, για παράδειγμα αυτά τα υπόλοιπα προς εκαθάριση στα ΕΕΛ είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα κοιτάξω να τονίσω ακόμα περισσότερο ε, σε αυτή τη γνωμοδότηση. Βέβαια είναι λίγο ε, στενά τα περιθώρια μας, δηλαδή δεν μπορούμε να αναφέρουμε πολλά σε ό,τι αφορά δηλαδή, το κείμενο, οπότε αναφερόμαστε μόνο σε ένα περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων. Υπάρχουν δηλαδή, αναφερόμαστε σε προγράμματα ε, για τα οποία χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και αν δεν υπάρχει αυτή η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Γι' αυτό και αναφέρουμε μόνο κάποια προγράμματα για τα οποία κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό. επίση το Horizon 2020 είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο πρέπει να γίνει μια καλύτερη διαχείριση των πόρων. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ε, πολλά στοιχεία για τα οποία στο πλαίσιο του ε, προγράμματος σχεδίου ε, Juncker μειώθηκαν εν είδη κονδυλίων και θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τέτοια κονδυλία για τον τομέα της εκπαίδευσης, της παιδείας και του πολιτισμού και αυτά από την πλευρά μου θα Περιμένω βέβαια έω τι 23 Μαρτίου του Ευχαριστούμε πολύ. Να αναφέρω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο επιπλέον ανησυχίε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα για τη Δημιουργική Ευρώπη και για το Erasmus Plus. Και δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει λίγο το πολιετές πλαίσιο και στα πλαίσια της αναθεώρησης αυτής θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Το έχουμε θίξει αυτό και στις συναντήσεις που είχαμε με τον Επίτροπο, νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον στη νέα προγραμματική περίοδο να δοθεί νέα έμφαση και μεγαλύτερη έμφαση στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα. 22 Μαρτίου 12 το μεσημέρι είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες. 26 Απριλίου θα ε, ψηφίσουμε εδώ πέρα και η αρμόδια επιτροπή τον Ιούνιο, ενώ θα πάει τον Ιούλιο η έκθεση αυτή στην ε, Ολομέλεια. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ πέρα και την κυρία Λούτσια Ρεκάλντε από το πρόγραμμα «Μέντια» καθώς επίσης και τον κύριο Μπάρκα και θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Είχαμε και τη δυνατότητα στο παρελθόν να θίξουμε τα ζητήματα τα οποία προβλέπονται σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και από τη Γενική Διεύθυνση Connect όσον αφορά το μηχανισμό εγγύσεων στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Έθιξα το ζήτημα των καθυστερήσεων. Χρειαζόμαστε βεβαιώσεις όχι μόνο προς το χρονοδιάγραμμα αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο νέος αυτός μηχανισμός εγγύσεων και δανειοδότησης. Ξέρετε ότι έχω κάνει πολλέ επίσημε και άτυπε επαφέ με εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μα την Επιτροπή να γνωρίζουμε πώ θα χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα στα πλαίσια του Δημιουργική Ευρώπη και πώς θα λειτουργήσει αυτός ο νέος μηχανισμός εγγύσεων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να ανταποκριθούν και οι ίδιοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί πέρα από τους υπόλοιπους εμπλεκομένους ε, φορείς σε εθνικό επίπεδο. Να καλωσορίσω λοιπόν τους δύο καλεσμένους μας και να δώσω το λόγο σε εσά. Έχετε συνολικά 15 λεπτά για να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τους συναδέλφους και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις ενδεχόμενες δικές σας απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας και μπορούμε να σας παρουσιάσουμε το πώς έχει κατάσταση ε, με το μηχανισμό εγγυήσεων για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Έχουμε έρθει εδώ λοιπόν για να σας κάνουμε μια ε, κοινή παρουσίαση με τη Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια. Να σας πω ποιο είναι το νομικό πλαίσιο, γιατί αυτός ο μηχανισμός αποτελεί έναν απόσπαστο κομμάτι του προγράμματος Creative Europe, την Δημιουργική Ευρώπη, που είναι όχι, που έχει ως στόχος καταρχήν την ε, διαφορετικότητα αλλά και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Συγκεκριμένοι στόχοι είναι καταρχήν και αναφέρουμε στους πρώτους δύο από αυτούς οι οποίοι ε, στηρίζουν το όλο εγχείρημα που είναι η ενδυνάμωση της οικονομικής δύναμης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ένα βιώσιμο τρόπο και δεύτερον να προωθήσουν την καινοτομία και τη διαχείριση της επιχειρηματικότητας. Προφανώς λοιπόν το εγχείρημα αυτό ε, και ο μηχανισμός αυτός σίγουρα στηρίζουν τα όσα έχουμε θέσει ως στόχους στο Creative Europe. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά να υπογραμμίσω πως πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό εγγύησεων και γι' αυτό έγιναν ε, ευρύτατες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή ε, κάποιες ενώσεις media, κάποιους φορείς, ε, συμβούλους, consultants και πρέπει να σας πω πως έχουμε ε, αποσπάσει από όλους αυτούς πολύ στεναρά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της συνέχισης αυτού του μηχανισμού. Είναι ένα μοναδικό ένας μοναδικός μηχανισμός που αποτελείται από δύο στοιχεία κλειδιά Καταρχήν κάνει το capacity building, την ε, οικοδόμηση δυναμικού, γιατί οι κλάδοι αυτοί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα ε, στη στιγμή της εξέβρεσης χρηματοδότησης. Πολλές φορές τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν κατανοούν τα βασικά τους στοιχεία και το πώς λειτουργούν αυτοί οι κλάδοι. Άρα λοιπόν με το capacity building θέλουμε να προσφέρουμε πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να αυξήσουμε ε, την κατανόηση που υπάρχει για τις ιδιαιτερότητες του κλάδου κάπως δηλαδή μέσω οικονομικών διαμεσολαβητών έτσι να μας δείτε και επίσης για την πρόσβαση της χρηματοδότησης, την πρόσβαση της χρηματοδότησης από μικρομεσαίες μέσω κάποιων εγγύσεων και αντεγγύσεων. Will make SMEs and the loans να σας πω λοιπόν πως υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, τα οποία καταστούν επιλέξιμες αυτές οι μικρομεσαίες. Πρώτο κριτήριο επιλεξιμότητας. Η μικρομεσαία αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να είναι επιχείρηση ε, του συγκεκριμένου κλάδου. Δηλαδή να εμπίπτει στο πεδίο του ορισμού του τι είναι δημιουργικούς ή πολιτιστικός κλάδος που είναι αυτός που περιγράφεται στη νομική μας βάση. Στον κανονισμό Creative Europe. Και βεβαίως εκεί θα πρέπει να είμαστε πάντα συνεπείς. Βλέπετε λοιπόν πως έτσι καλύπτουμε μια μεγάλη γκάμα κλάδων, αρχιτεκτονικά, οπτικοακουστικά, φεστιβάλ, λογοτεχνία, μουσική, τεράστιο το πεδίο εφαρμογή. Δεν θα απορριθμίσω καθέναν που εντάσσεται σε αυτό. Επίσης, μικρομέσαια, μικρομέσαια. Εδώ έχουμε δύο πλήρους ε, ορισμούς του τι είναι μικρομεσαία. Πρώτα απ' όλα είναι ο ορισμός που έχουμε στην νομική βάση του Creative Europe και τονίζω πως καλύπτει όχι μόνο τις μέσες επιχειρήσεις αλλά και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης προσθέσαμε εδώ επιχειρήσεις που είναι μικρομεσαίες, μόνο μικρές και μόνο μεσαίες και που δεν εμπίπτουν ακριβώς ε, σε αυτόν τον ορισμό γιατί οι μετοχές τους ανήκουν σε δημόσιους ε, φορείς και αυτό επιτρέπει σε ιδρύματα όπως τα θέατρα, τα διάφορα ιδρύματα να είναι επίσης επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού. Άρα λοιπόν έχουμε διευρύνει εδώ το πεδίο μας. Μουσεία επίσης. Αρκεί να ε, καλύπτουν και τα υπόλοιπα κριτήρια. Για τα δάνεια, για τα δάνεια λοιπόν. Ο, κλάδι, ο κλάδος αυτός πολύ δύσκολα βρίσκει χρηματοδότηση και πολλές φορές τα ε, χρηματοδοτικά ιδρύματα ζητούν για προσωπικές εγγύησεις. Οπότε εδώ μέσω αυτού του μηχανισμού δεν χρειάζονται ε, εγγυήσεις υλικέ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν μπορούν να ζητήσουν το δάνειό σου, το στεγαστικό ως εγγύηση. Αντίθετα, τα χρηματοπιστικά ιδρύματα θα ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν τα άειλα ε, ε, περιουσιακά στοιχεία των ε, εταιριών ως εγγύηση και αυτό θα φέρει μια αλλαγή στη δανειστική πολιτική αυτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Άρα λοιπόν μπορούμε να καλύπτουμε άειλα και άλλα στοιχεία ενεργητικού και επίσης να φτάνουν σε ένα μέγιστο 10 εκατομμυρίων ευρώ ανά δάνειο. Αυτά ως προς τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Τώρα, να σας πω πως θα προσφέρουμε και πραγματογνωμοσύνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή γιατί όπως σας εξήγησα καλύπτουμε και τις δύο όψεις ε, του φάσματος θα είμαστε ανοιχτοί σε χρηματοπιστωτικού για μεσολαβητέ, όχι σε ιδρύματα απευθεία, με σκοπό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μπορούν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο του να δανείζουν χρήματα στο συγκεκριμένο αυτό κλάδο. Δηλαδή θα μιλάμε για μια πολύ ε, κοντινή προσπάθεια η οποία θα δημιουργήσει ε, capacity building στην πράξη. Είναι hands-on αυτή και πολύ στοχευμένη η προσέγγιση ε, τουλάχιστον ε, στα δάνεια τα οποία θα αποφασιστεί να χορηγηθούν. Τι έχουμε λοιπόν συμφωνήσει με το ΑΕΦ να έχουμε καταρχήν να κάνουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης που θα καλύψει και την πλευρά της ζήτησης και την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή χρηματοσυντητικά ιδρύματα φαινός και τον ε, κλάδο το δημιουργικό και το πολιτιστικό. Άρα λοιπόν ο μηχανισμός θα ε, ε, ασχοληθεί με, τους, ε, με τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και εμείς από την πλευρά μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνουμε την εκστρατεία ενημέρωσης έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι παίκτες στους κλάδους να γνωρίζουν πως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αυτή η χρηματοπιστωτική ενδιάμεση θα πρέπει να προσφέρουν επιχειρηματικό σχέδιο ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει να αποδεικνύουν πως υπάρχει και συστράτευση και πολύ ε, ε, στοχευμένη προσέγγιση των επιχειρήσεων για να του επιτρέψουμε να εισέλθουν στο πρόγραμμα. Να παρουσιάσω κάποιες από τις δράσεις που σκοπεύουμε να λάβουμε και σε επίπεδο εκδηλώσεων και περιεχομένου. Λοιπόν, εκδηλώσεις στα κράτη-μέλη, εκεί θα χρησιμοποιήσουμε ε, το Media Desk για το Creative Europe που υπάρχει όχι μόνο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις συνδεδεμένες χώρες ως πολλαπλασιαστές που θα χρησιμοποιήσουν και το Ευρωπαϊκό Βήμα ε, Ταινιών, το European Film Forum, ως τόπο διάδοσης ε, πληροφοριών. Θα παρουσιάσουμε φυλάδια, ε, ε, ενημερωτικά τεύχη, μπροσούρες στο site μας και στο Access to Finance και στη σελίδα εκεί θα έχουμε τις προφορίες αυτές έτσι ώστε να πλησιάσουμε στον δυνατόν περισσότερο. Σε αυτή τη στιγμή Έχουμε την συμφωνία εξουσιοδότηση, η οποία έχει συμφωνήσει στα περισσότερα σημεία, θα ξεκινήσουν οι εσωτερικέ διαδικασίε να τρέχουν σύντομα και ελπίζουμε πω η συμφωνία αυτή ε, θα υπογραφεί γύρω στο Μάιο. Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για να μην χαθεί καθόλου χρόνος μετά την υπογραφή θα στέλνουν τι αιτήσει του οι τράπεζε και κάποια χρηματοπιστικά ιδρύματα ενδεχομένω να έχουν ήδη ε, επιλεγεί στο τρίτο τρίμηνο, δηλαδή στο δεύτερο εξάμεινο τη φετινή χρονιά, έτσι ώστε μέχρι τα τέλη χρονιά να έχουμε κάτι στα σκαριά και στην αγορά. Οι εκστρατείε ενημέρωση θα αρχίσουν να τρέχουν αφού η συμφωνία υπογραφεί και καθ' όλη τη διάρκεια τη χρονιά. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί και παραμένουν ανοιχτοί μέχρι το 2020, οι προσκλήσει δηλαδή για τους διαγωνισμούς, οπότε θα είναι μια ε, συνεχής διαδικασία. Για να ανακεφαλαιώσω, έχουμε αυτή τη δυτή ε, στόχευση που είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση ε, η οποία θα προσπαθεί να δώσει δάνεια σε μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον πολιτιστικό και ε, στον κλάδο χωρίς να χρειάζεται η εταιρεία που δανείζεται να καταθέσει την προσωπική της περιουσία ως εγγύηση. Μέχρι το 2020 ξέρετε ποιος είναι ο προϋπολογισμός, είναι 120 εκατομμύρια και νομίζω ότι αυτό θα αμοχλεύσει γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην αγορά. Συμμετοχή για όλα τα κράτη-μέλη, όπως επίσης και για τις χώρες ε, ΕΟΧ, όχι στις συνδεδεμένες χώρες. Και η εφαρμογή, όπως σας είπα, κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για να ε, ξεπεράσουμε τις καθυστερήσεις και να προχωρήσουμε σε εφαρμογή το 2016 ήδη. Um, <clears throat> ε, πολύ σύντομα από την πλευρά πολιτισμού να προσθέσω κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε συνεργαστεί εντατικά με την Γενική Διεύθυνση Connect κάτω τους τελευταίους μήνες και έχουμε φροντίσει οι φάκελοι οι οποίοι θα επιλεγούν για ε, χρηματοδότηση από τα τραπεζικά ιδρύματα θα είναι διαφοροποιημένοι μεταξύ τους και θα υπάρχουν και οι κατάλληλες διατάξεις που θα ισχύουν και βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των διαφόρων τομέων για αυτό τον ε, μηχανισμό ε, παροχής εγγυήσεων και, θεωρού, και είμαστε πεπισμένοι ότι ε, λίγους μήνες μετά από την ε, έναρξη αυτού του προγράμματος, ε, μετά από, δηλαδή από την επιλογή των πρώτων project και την συμμετοχή των πρώτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα δούμε ότι θα αρχίσουν να αποφέρουν καρπούς αυτά τα μέτρα, δηλαδή δημιουργίας περισσότερης εμπιστοσύνης και εμπιστοσύνης δηλαδή για χρηματοδότηση από την πλευρά του τραπεζικού τομέα προ τον ε, τομέα του πολιτισμού, τον κλάδο του πολιτισμού και τη ε, δημιουργία. Και ε, κάτι τέτοιο βέβαια είναι ένα από του βασικού στόχου του προγράμματο Δημιουργική Ευρώπη, δηλαδή που διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Δηλαδή ότι ε, έχουμε το συνδυασμό των ε, υφιστάμενων μέτρων με πιο μακροπρόθεσμα μέτρα ακριβώ χρηματοδότηση ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα πολιτισμού και τη δημιουργία. Έτσι διασφαλίζουμε δηλαδή ότι από τώρα έως το 2020 τα η ενίσχυση η οποία παρέχεται στα κράτη-μέλη σε τέτοιου είδου μικρομεσαίε επιχειρήσει θα αποτελεί πλέον σε ένα συστατικό στοιχείο ε, του, του και έτσι θα καταφέρουμε να κλείσουμε και αυτό το κενό που υπάρχει στο επίπεδο της χρηματοδότησης. Η επικοινωνία σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή ε, πολλοί φορείς ε, στον τομέα του πολιτισμού γνωρίζουν ότι ε, έρχεται αυτό το πρόγραμμα και θα εστιάσουμε βέβαια τις προσπάθειες μας για επικοινωνία, για προβολή στα κράτη-μέλη εκείνα όπου θα ξεκινήσει και βέβαια θα διευρύνουμε αυτές τις ε, προσπάθειες ε, και στο μέλλον. Και αυτό βέβαια το διασφαλίζουμε και μέσω της συμμετοχής όλων των δικτύων και όλων των μεγάλων φορέων οι οποίοι συμμετέχουν και είναι πάντοτε η βασική μας εταίροι στο επίπεδο των πρωτοβουλειών χρηματοδότησης έτσι ώστε να μπορέσουμε πράγματι να εφαρμόσουμε στην, και να μεταφέρουμε αν θέλετε στην πραγματικότητα του κλάδου του πολιτισμού αυτόν τον μηχανισμό. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνοπτική αυτή παρουσίαση, πάρα πολύ σαφής όμως. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε να θέσουμε φαντάζομαι κάποια ερωτήματα για να καταφέρουμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που είχαν ζητήσει το λόγο. Πρώτη η κυρία Έλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Χρειάστηκε πολύ χρόνο μέχρι να έχουμε την πρότασή σας, οπότε είναι λίγο κρίμα που δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Όμως ελπίζω πως τώρα με τα κονδύλια και με τη μόχλευση των 600 εκατομμυρίων ευρώ θα βοηθηθεί ο κλάδος. Για τον ίδιο τον κλάδο να σας πω πως έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Εάν θυμηθούμε τη νομική βάση και τα όσα συζητήσαμε για το πρόγραμμα Creative Europe, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο πως δεν θέλαμε μόνο να καλύψουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά να συμπεριλάβουμε και τα μικρά ε, καλλιτεχνικά project, πολιτικά project. Οπότε ε, θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση. Είναι ανοιχτέ οι προσκλήσει αυτέ και για τέτοιου είδου μικρά πολιτιστικά project, γιατί αν θέλει κανεί που τι τρέχουσε συνθήκε να ανοίξει σε project που έχουν να κάνουν με την ενσωμάτωση των προσφύγων, ή με τον διαπολιτισμικό διάλογο για να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση ε, του πολίτη ότι ανήκει ε, τότε θα πρέπει να γίνει και κάτι τέτοιο. Επιτρέπεται λοιπόν γιατί μέχρι στιγμής είπατε έχει ανοίξει σε μικρές επιχειρήσεις οι εταιρείε. Δεν ξέρω λοιπόν τι γίνεται με τα project, με τα έργα τα οποία δεν ε, είναι εμπορικά, αλλά είναι μη εμπορική φύση, γιατί το είχαμε συζητήσει και στα πλαίσια του προγράμματο και θα ήθελα να μου απαντήσετε. Πείτε μου, για να είμαι βέβαιη πως σε πολιτικό επίπεδο μπορούμε να πούμε πως τα μικρά πολιτικά project καλύπτονται από αυτό το μηχανισμό. Ε, Ευχαριστούμε. Στρογεύσκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο από το ότι καταρχάς ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό. Καλύπτει ένα τεράστιο κενό και νομίζω ότι θα πρέπει μέσω του προγράμματος αυτού να επενδυθούν περισσότερα χρήματα στον τομέα του πολιτισμού. Σε καμία περίπτωση δεν κατασπαταλάμε χρήματα όταν μιλάμε για πολιτισμό. Ο πολιτισμός ίσως να μην με επένδυση. Θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις τώρα σε σχέση με την παρουσίασή σας. Αυτές οι διαφορετικές κατηγορίες που μας παρουσιάσατε, τι είναι τελικά, είναι πιστώσεις, είναι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, δάνεια γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σύγχυση πολλές φορές στους χρήστες. Αν για παράδειγμα παίρνουμε ένα δάνειο, μια πίστοση, πρέπει κάποια στιγμή να το αποπληρώσουμε. Άλλα πράγματα όμως ισχύουν αν η χρηματοδότηση πάρει τη μορφή επιδότησης ή οικονομικής ενίσχυσης. Επίση, το ίδιο ισχύει και για τα επιτόκια. Διαφορετικά τα επιτόκια όταν μιλάμε για δάνειο ή δεν υφίστανται καθόλου επιτόκια όταν μιλάμε για επιδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω καλύτερα πώ λειτουργεί ο μηχανισμό αυτό στις διαφορετικέ κατηγορίε, τι οποίε παραθέσατε. Τι σημαίνει επένδυση 120 εκατομμυρίων ευρώ με τον ένα τον άλλο τρόπο και πώς θα ανανεωθεί επίσης το ταμείο αυτό εφόσον προβλέπετε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Τζιμπράσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το δικό μου το ερώτημα ομοιάζει με αυτό το οποίο έθεσε ο συνάδελφος πριν από λίγο. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για να ενισχύσουμε κάποιους συλλόγους, κάποιες καλλιτεχνικές πολιτιστικές ενώσεις, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, δεν λειτουργούν με τρόπο κερδοσκοπικό πάντα, δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στους συλλόγους αυτούς τους οργανισμούς. Α, Λουίτζι Μόργανο, συγγνώμη, δεν σε είχα δει. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με την παρουσίαση αυτή και πραγματικά ανταποκρίνει το μηχανισμό αυτό σε μια τεράστια ανάγκη που είχε εντοπιστεί στον τομέα. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να γνωρίζω αν προβλέπετε κάποια κριτήρια προτεραιότητας όσον αφορά την ανάθεση αυτής της χρηματοδότησης. Δεύτερον, σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε πάλι εδώ πέρα να θέσουμε πολλά ερωτήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξολογήσετε περισσότερο πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό σε σχέση με τις τράπεζες. Λέτε ότι οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί θα πρέπει να καταδείξουν ότι έχουν ε, ήδη υποστηρίξει ανάλογα σχέδια στο παρελθόν. Σε τι ακριβώς αναφέρεστε όταν λέτε κάτι τέτοιο, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ετέθησαν διάφορα ερωτήματα. Να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά τον κανονισμό για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Ξέρουμε ότι κάποιες διατάξεις ήταν κάπως γενικέ. γενικές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Το ζήτημα των εγγυήσεων, του μηχανισμού αυτοεγγυήσεων. Όπως λέτε εσείς να απευθύνεστε μόνο σε τράπεζες, αλλά απευθύνεστε και σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Υπάρχουν ήδη κάποιοι τέτοιοι οργανισμοί σε ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία μπορούν να καλύπτουν και εγγύησει ή μπορεί σε ορισμένου από αυτού να υπάρχει απαραίτητη πυρογνωμοσύνη όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού. Σε σχέση με αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι πριν από λίγο, να θέσω την εξή ερώτηση. Πώς θα καταφέρετε να επιλέξετε κάποιους εμπειρογνώμονες για το ζήτημα του capability. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, έχετε επιλέξει αυτούς του εμπειρογνώμονες για την οικοδόμηση αυτή των ικανοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια των κριτηρίων, όπως είπε και ο Λουίς Μόργανο, να καταφέρουμε να, έχουμε δύο κατηγορίες, όχι μόνο το ότι όχι ένα κριτήριο που θα έχει να κάνει μόνο με τον πολιτισμικό εκπαιδευτικό τομέα, αλλά θα πρέπει να έχουμε και εταιρείε ή οργανισμούς non-profit, μη κερδοσκοπικούς. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να δώσουμε μια ευκαιρία και σε αυτούς τους συλλόγους πολλές φορές μπορεί να είναι ακόμα και μουσεία. Αν αφήσουμε εκτός αυτές τις, αυτούς τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, απευθυνόμαστε μόνο σε εταιρείε και σε επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν και οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί να μπορούν να καλύπτουν εγγυητικά αυτούς τους οργανισμούς. Πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο δανειοδοτικό που να καλύπτει αυτούς αυτές τις πολύ διαφορετικές μορφές ε, οργανισμών, εταιριών, επιχειρήσεων κτλ. Προσπαθούμε επίσης να καλύψουμε εμείς διάφορους τομείς εδώ πέρα, αλλά προσπαθούμε να έχουμε και μία γεωγραφική κάλυψη. Προβλέπετε αυτό στη δική σας την αξιολόγηση. Φαντάζομαι ότι θα επιλέξετε τους καλύτερους, αλλά παρόλα αυτά έχετε δώσει μια κάποια, ένα κάποιο κίνητρο προς τους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς να προχωρήσουν σε μια ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη των ε, επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτήσουν. Επίσης, ε, βρισκόμαστε ήδη ή θα φτάσουμε στα μέσα του 2016 σύντομα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία ανοιχτή προκήρυξη. Να μην προχωρήσουμε δηλαδή σε πολλές επιμέρους κατακαιρματισμένες προκήρυξεις, αλλά να έχουμε τουλάχιστον από τα μέσα του 2016 και μετά μία ανοιχτή προκήρυξη και μπορείτε αυτή τη στιγμή να αποστικοποιήσετε κάπως τον αριθμό των χρηματοδοτικών οργανισμών πιστεύετε ότι θα ανταποκριθούν στην πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ. Well, thank you. I will go through the different questions. Θα τα πω ε, ένα-ένα. Τώρα, την ερώτηση που έγινε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Why I will repeat it is that um, under the definition of SMEs is not only medium-sized enterprises. Λοιπόν, δεν είμαστε περιορισμένοι μόνο σε μικρές, πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις ε, και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε Συγγνώμη, ε, διορθώνει ή ε, καλύπτουμε μόνο μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης και μεσαίες επιχειρήσεις. Ε, αυτά περί τη κάλυψη. Τώρα για τα μη κερδοσκοπικά project. Όταν συζητήσαμε την επιλεξιμότητα των ε, ε μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είπαμε μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε κάποιες επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές ανήκουν σε δημόσιους φορείς. Για παράδειγμα, ιδρύματα, μουσεία, έτσι ώστε και αυτά να έχουν πρόσβαση χρηματοδότηση παρόλο που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Είναι ξεκάθαρο πως αυτή είναι ε, μια δυνατότητα που υπάρχει, αλλά ο μηχανισμός μας είναι μηχανισμός αγοράς. Αυτό μην το ξεχνάμε. Η βιωσιμότητα δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλίζεται στην αγορά. Τώρα, οι μικρές, πολύ μικρές και μεσές επιχειρήσει, βεβαίω και καλύπτονται σύμφωνα με τον ορισμό που παρουσίασα στην αρχή. για το χαρτοφυλάκιο και την ερώτηση που έγινε σχετικά. Ο μηχανισμός αυτός ακολουθεί ε, την προσέγγιση διαχείριση χαρτοφυλακίου, δηλαδή τα χρηματοψηφικά ιδρύματα που θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το μηχανισμό εγγύησεων θα καταφθάνουν με ένα χαρτοφυλάκιο και ε, θα κοιτάμε και το κατά πόσο διαφοροποιημένο αυτό το χαρτοφυλάκιο τη στιγμή της αξιολόγησης. Θα υπάρχει λοιπόν μια εγγύηση της τάξης του μέχρι 70% ε, αναδάνειο και ένα 25% που θα χορηγείται με βάση το χαρτοφυλάκιο. Άρα λοιπόν το χαρτοφυλάκιο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του μηχανισμού γιατί στο χαρτοφυλάκιο θα μπορούμε να έχουμε ένα συνδυασμό διαφόρων κλάδων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σχήμα το οποίο θα είναι πολύ πιο διαφοροποιημένο με πολύ μεγαλύτερη εκπροσώπηση αυτών των ε, κλάδων. Γιατί η γεωγραφική κάλυψη εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ποσά τα οποία θα είναι διαθέσιμα. Δηλαδή όσο πιο πολλά χρήματα έχει κανείς, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες να καλύψουν μια μεγαλύτερη γκάμα χωρών. Αυτή τη στιγμή με τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα έχουμε υπολογίσει πως θα μπορούσαμε να καλύψουμε γύρω στα τέσσερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό ως απάντηση. Αλλά όπως είπα υπάρχουν περιορισμοί που σε αυτή τη φάση δεν μας επιτρέπουν να καλύψουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό χώρων ή χρηματοπιστικών ιδρυμάτων. Για την επιλογή των ε, εμπειρογνωμόνων που θα βοηθήσουν στο capacity building να σας πω πως και εδώ θα δημοσιευθεί πρόσκληση που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ε, υπογραφή της Συμφωνίας Εξουσιοδότησης και ποιοι θα είναι αυτοί οι εμπειρογνώμονες. Μπορεί να είναι εκπρόσωποι του κλάδου, μπορεί να είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορεί να είναι consultants. Ακόμα το θέμα αυτό το έχουμε αφήσει πάρα πολύ ανοιχτό. Και θα έχουμε και κάποιον ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό όλων των εμπειρογνωμόνων ε, του capacity building. Και όλα αυτά θα λάβουν υπόψη και τα γεωγραφικά στοιχεία αλλά και τις ιδιωτερότητες των κλάδων. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να κινητοποιηθούν πάρα πολλοί εμπειρογνώμονες στα πλαίσια του capacity building. Αν ξεκινήσει λοιπόν η πρόσκληση αφού αμέσως μετά την υπογραφή του, της συμφωνίας το δεύτερο εξάμεινο του 2016 και πριν το τέλος χρονιάς σίγουρα θα έχουμε κάτι που να λειτουργεί. I think I have... Uh, would you like to add Θέλεις να προσθέσεις κάτι, ναι, στα γρήγορα. Μια τράπεζα συνήθως η οποία θα επιλεγεί και μετά θα συνάψει σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και αυτής θα, θα ξεκινήσει επιλέγοντας φορείς, ε, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ε, οργανισμούς πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, νομικούς φορείς, δημοσίου δικαίου, και δεν θα ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία για τη δανειοδότηση ενός project. Αντίθετα, αυτό που θα γίνει εδώ είναι να έχουμε φορείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα σε τέτοιου είδους χρηματοδότηση μέσω project γιατί αν δεν έχει κανείς project δεν θα μπορεί να λάβει δάνειο. Για να συνδυάσουμε έτσι τις διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης, νομίζω πως εδώ αυτό το οποίο στείλουμε είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι σήμερα. Έχεις λοιπόν τις, ε, τα κριτήρια επιλογής, τη νομική βάση, το ποιοι είναι οι στοχευμένοι φορείς ε, αυτού του κλάδου στην Ευρώπη που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έχει και τους υπόλοιπους στα πολιτικά στα μίντια. Εδώ λοιπόν ανοίγουμε στις μικρομεσίες, στις πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις και ε, στις μικρομεσίες επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως επίσης και στους ε, φορείς οι οποίοι είναι οι μη έτσι ώστε να έχουν εγγυημένες δυνατότητες να δανειστούν από τις τράπεζες. Οπότε δεν έχει να κάνει με τις επιχορηγήσεις που προσφέρει συνήθως ε, η Creative, το πρόγραμμα Creative Europe. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι μηχανισμός που εξασφαλίζει εγγύησεις. Να σας υπενθυμίσω δε πως αυτός ο μηχανισμός προσφέρει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να ανοίξει ε, κατευθείαν στα χρηματοπιστικά ιδρύματα αλλά και κατευθείαν σε μικροεπιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά μέσω των αντικοιήσεων θα μπορούσαν να έχουμε και συνδυασμό χαρτοφυλακίων μεταξύ χρηματοπιστικών ιδρυμάτων έτσι ώστε να καλύψουμε και τους πάρα πολύ μικρού μεγέθους ε, φορείς. Κυρία Τρούπελ και μετά εγώ. Sorry for insisting, but I really would like to ask back. Um... Ζητώ συγγνώμη που επιμένω, αλλά θα ήθελα να τονίσω μια πτυχή. Άκουσα ήδη κάτι πρόταση, πρώτα ομιλία που αναφερθήκατε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές οδοντές, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι σε πολλά κράτη-μέλη, ειδικότερα στη δική μου χώρα, στη Γερμανία, υπάρχουν κάποια προγράμματα ε, στον τομέα του πολιτισμού που είναι σε κάποιο ε, μέχρι βαθμό αυτόνομα, δηλαδή ε, είναι ένα πρόγραμμα πολιτισμικού χαρακτήρα το οποίο απευθύνεται γενικότερα σε φορείς στον χώρο του πολιτισμού. Οπότε ε, θα ήταν, ε, θα μπορούσε να ενταχθεί, να είναι τέτοιου είδους προγράμματα επιλέξιμα στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυήσεών σας νομίζω πως θα πρέπει να εξετάσουμε επακριβώς ποια είναι, ποιο είναι το είδος αυτών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Σας είπα ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας. Για παράδειγμα θα πρέπει να είναι μικρομεσαία επιχείρηση και προσπαθήσαμε να διευρύνουμε όσο γίνεται περισσότερα αυτόν τον ε, ορισμό. Γιατί αυτό που αναφέρεται αυτή τη στιγμή ως ορισμός ε, στον ε, κανονισμό για τη Δημιουργική Ευρώπη αναφερόταν μόνο σε μικρέ, πολύ μικρέ επιχειρήσει. Αλλά εμεί τώρα προσπαθήσαμε να διευρύνουμε αυτόν τον ορισμό για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερε επιχειρήσει από τον χώρο του πολιτισμού. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να τηρήσουμε τα όρια που μα θέτει αυτό ο ορισμό. Δηλαδή, ο ίδιο ορισμό τη ε, μικρομεσαία επιχειρήση που έχουμε θέσει αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητα. Ε, Ένα ακόμα ερώτημα. Είναι πολύ σημαντικά τα όσα είπατε για τι αντεγγύσει. Είπατε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εθνικές εγγύησεις, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αντεγγύησεις ως επιπλέον μηχανισμός. Όσον αφορά επίσης το ζήτημα της νομικής βάσης, είχε προκύψει στο παρελθόν το πρόβλημα αυτό, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώς ορίζεται ή ποια νομική βάση χρησιμοποιείται στα πλαίσια της συμφωνίας εξοδότησης, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των εγγύσεων. Εμείς στα πλαίσια του κανονισμού λέμε ότι δεν μπορούν να ζητηθούν προσωπικές εγγύησεις από τους φορείς. Ακριβώς επειδή ο κλάδος αυτός είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος, γιατί ε, πολύ συχνά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για, ένα, για πάρα πολλά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν οι πολιτιστικές αυτές εταιρείε, οι εταιρείε στον τομέα του πολιτισμού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέγαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να προβλέπεται ως εγγύηση και χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην πράξη, εσείς την προκήρυξη που θα κάνετε, πώς θα ορίσετε ακριβώς αυτή την έννοια, πώς ακριβώς θα αναφερθείτε στο ότι δεν υπάρχει υποχρέωση προσωπικών λεγόμενων εγγύσεων. Και σας το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι πολύ συχνά το ότι δυσκολεύονται οι εταιρείε αυτέ να πάρουν δάνεια χρηματοδότηση έχει να κάνει ακριβώ με το ότι δεν μπορούν όπω άλλε εταιρείε να προσφέρουν ω εγγύηση περιουσιακά υλικά στοιχεία. Αυτό προκύπτει ιδίω με τι τράπεζε ω πρόβλημα. Ευχαριστώ. Όπω είπατε κι εσεί, το στοιχείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στα πλαίσια τη συμφωνία εξοδότηση το έχω αποσαφηνίσει και στα πλαίσια τη καμπάνια ενημέρωση που θα κάνουμε θα το αποσαφηνίσουμε περαιτέρω. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά και κρίσιμα στοιχεία του μηχανισμού αυτού εγγύσεων. Κύριος έχει το λόγο. Κατάλαβα τα όσα είπατε για τις εγγύησεις. Από την άλλη αναφερθήκαμε και σε άλλες πιστώσεις, σε δάνεια, σε επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι διαφορετικοί όροι, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για δάνεια αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα χρήματα τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν. Διαφορετικά πράγματα όμως ισχύουν όσον αφορά άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικής υποστήριξης όπως οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις κτλ. Μπορείτε να μας δώσετε και προς αυτό μια απάντηση, γιατί αυτό θα μπορούσε να πειράσει ιδιαίτερα τις δυνατότητες δανειοδότησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Um, Αυτό θα ακολουθήσει τις συνηθισμένες εμπορικές πρακτικές, εάν καταλάβω την ερώτησή σας. Άρα λοιπόν θα τοποθετηθούν ως προϊόντα στην αγορά τραπεζικά προϊόντα τα οποία θα προστατεύονται λόγω της χρήσης του μηχανισμού, του εγγυητικού μηχανισμού. Οπότε θα βγαίνουν στην αγορά στους τραπεζικά προϊόντα και θα ακολουθούν τη συνήθεια εμπορική πρακτική, εάν απαντώ σωστά. Ci sono altre questioni. Άλλες ερωτήσει. Λοιπόν, πολύπλοκο το ζήτημα, το βλέπουμε όλοι, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα μηχανισμό εγγύσεων, για ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα δοκιμάσουμε βασικά στο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θελήσαμε στα πλαίσια του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη να έχουμε ένα μηχανισμό χρηματοδότησης που να φωτίζει με διαφορετικό τρόπο το ζήτημα της δανειοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καταφέρουμε δηλαδή με έναν τρόπο καινοτόμο να χρηματοδοτήσουμε έναν κλάδο ο οποίο δύσκολα χρηματοδοτείται στο παρελθόν. Τίθεται το ζήτημα αυτό των πολύ μικρών επιχειρήσεων Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουν να συμμετάσχουν, όπως είπατε, και πολλές άλλες εταιρείες, δηλαδή φορείς, ιδρύματα και όχι μόνο επιχειρήσεις. Και το σημαντικότερο είναι να μην καταλήξουμε σε ένα κατακαιρματισμένο περιβάλλον με 28 διαφορετικές δυνατότητες χρηματοδότησης, αλλά να έχουμε έναν ενιαίο μηχανισμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες παρουσιάζονται από τη μία χώρα στην άλλη και να καταφέρουμε δηλαδή να κάνουμε κάποια προγράμματα επιλέξιμα για το μηχανισμό αυτό, τα οποία όμως να μην επικεντρώνονται στις συγκεκριμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στο Νότο για παράδειγμα ή μόνο στο Βορρά. Θα πρέπει να μπορούν και άλλοι φορείς πέρα από τις εταιρείες ή τις επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στην αγορά με έναν εντελώ εμπορικό προφίλ να μπορούν να χρηματοδοτούνται από το μηχανισμό αυτό. Θα θέλαμε κι εμείς ε, ή δυνατόν να έχουμε αυτή τη συμφωνία εξοδότησης όταν αυτή εγκριθεί και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε και αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης, αυτή την εκστρατεία ενημέρωση Πολλοί συναδελφοί και από τη δική μου τη χώρα έχουν πει ότι δεν υπάρχουν ακόμη απαραίτητες πληροφορίες. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στα πλαίσια μιας ενημερωτικής εκστρατείας να εμπλακεί περισσότερο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικής Ανάπτυξης ή για πολλά άλλα προγράμματα. Να καταφέρουμε να έχουμε δηλαδή έναν καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου από κοινού να μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την εκστρατεία ενημέρωση. ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θεσιμότητά σα. ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και ή δυνατόν μόλις ε, καταφέρετε να έχετε περισσότερες και